Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ, γιατί θα αρχίσει αμέσω η συνεδρία τη Επιτροπή μας. Καλησπέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Επαναλαμβάνω, άρχεται η συνεδρίαση. Σημείο πρώτο της ημέρησης διάταξης, ψηφοφορίες. Καταρχήν για τον προϋπολογισμό του 2017. Ε, έχουμε και ένα τηλεοπτικό συνεργείο που θα μαγνητοσκοπήσει τη συνεδρίαση το απόγευμα. Εξού και η καμεραμάν που βλέπετε στην αίθουσα. Θα γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ, γι' αυτό και θέλουν να μαγνητοσκοπήσουν μερικά στιγμιότυπα από τη συνεδρίασή μας. Μία μόνο ψηφοφορία έχουμε σήμερα και αφορά τον προπολογισμό του 2017. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Νταντσίλα. Δεν ξέρω αν θα θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους ε, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της γνωμοδότησής μου και να ευχαριστήσω επίσης και τη γραμματεία. Ευελπιστώ ότι εκπονήσαμε μια καλή γνωμοδότηση που θα υπερψηφιστεί και εδώ και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Νταντσίλα. Οπότε περνάμε στη ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 δεν θα την ψηφίσουμε για την εγγλωσσική 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Μάλιστα, ναι. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 9. Μια στιγμή να ρυθμίσουμε εδώ το μηχάνημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Mm 17 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ, καμία ψηφοκατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Νταντσίλα. so Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης θέμα ο ρόλος των γυναικών στην επίλυση διαφορών και στην συμφιλίωση.

Ε, για τις τέσσερις ε, περιμένουμε τους καλεσμένους μας, τους εμπειρογνώμονες. Οπότε μας έχει απομείνει ένα τέταρτο. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς τους καλεσμένους μας. Στις τέσσερις λοιπόν θα καταφτάσουν οι καλεσμένοι μας και μέχρι τότε θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.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

Bueno, queridos colegas. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Περνάμε στο σημείο που αφορά το ρόλο των γυναικών στην επίλυση των συγκρούσεων και τη συμφιλίωση. Θα κάνω μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Σουμάχερ της UN Women. Τη γνωρίζουμε την κυρία Σουμάχερ. Είχαμε την χαρά να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί της πολλές φορές. Την ευχαριστούμε και πάλι που ξανά ήρθε στην ε, Επιτροπή μας για να λάβει μέρος αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Και επίσης έχουμε την κυρία Ράμπι Ντεμαελίν και τον κύριο Βασάν Αραμίν από τον κύκλο γονέων Parent Circle που είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που απαρτίζεται από οικίους Παλαιστινίων και Ισραηλινών που έχασαν συγγενείς τους στη σύγκρουση και αποφάσισαν να συνεργαστούν για την εδραίωση της ειρήνης και τη συμφιλίωση. Είναι πραγματικά αξιέπαινο και καταπληκτικό το έργο τους, το έργο αυτής της οργάνωσης που είναι οργάνωση κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τέτοιε κοινωνικέ και πολιτικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να του ευχαριστήσω θερμά και για την παρουσία του εδώ, αλλά και για την προσπάθεια που κάνουν, τον αγώνα που δίνουν καθημερινά στην οργάνωσή τους. Και στις 6 το απόγευμα όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της ε, Επιτροπής μας θα έχουμε και τα εγγένεια μιας έκθεσης φωτογραφίας με συνδιοργάνωση από το Parent Circle Families Forum από αυτές τις πενθούσες οικογένειες Ισραηλινών και Παλαιστινίων που συμμετέχουν σε αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση και είστε προσκεκλημένοι όλοι και όλες σε αυτή την έκθεση φωτογραφίες και στα εγγένεια που θα γίνουν στις 6. Θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας. Πρώτα όμως ε, θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο της εκστρατείας ε, «Κάντε βήματα για την ειρήνη». Είναι έτοιμο το βίντεο για να το προβάλλουμε. Ε. Δεν προβλέπετε διερμηνία για το βίντεο. Ναι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 Σίγουρα μας άγγιξε αυτό το βίντεο. Και επιβεβαίωσε την προσήλωσή μας ε, σε αυτό το έργο. Ο καθένας μας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του σε αυτή την προσπάθεια για την ανέβρεση της λύσης και την εδραίωση της ειρήνης και την επίτευξη της συμφιλίωσης. Αυτό που επιδιώκουν ε, και οι οικογένειες αυτές που παρά το πένθος τους συμμετέχουν σε αυτή την οργάνωση προσπαθώντας και δουλεύοντας για τη συμφιλίωση. Θα περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην Ρόμπι Ντάμελη για 10 λεπτά περίπου, ώστε να μείνει κάποιος χρόνος για τη συζήτηση. Η κυρία Ντάμελεν. Yeah. So actually in the interests of gender equality... φιλοσοφίας. Ξέρετε ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κρατάει το όπλο τον οποίο τον στοχεύει. Δεν ξέρουμε. Και όπως όλοι οι Ισραηλοί πήγε να κάνει την θητεία του έφεδρος και βεβαίως δεν ήξερε κανείς ότι θα βρεθεί στα κατεχιόμενα. Αυτό που μου είπε βέβαια ήταν ότι αν δεν πάω τι θα γίνει με τους φοιτητές μου. Οι φοιτητές ε, και εκείνοι έτσι κι αλλιώς ε, θα συμμετείχαν στον Ισραηλινό στρατό και αυτό που σας είπα και πριν είναι πολύ σημαντικό ότι κανείς δεν ξέρει ποιος είναι πίσω από ένα όπλο. Και βεβαίως ακριβώς το ίδιο που να πούμε και για τους νέους Παλαιστίνιους. Ένας νέος ο οποίος σπουδάζει φιλοσοφία, ο οποίος θα πήγαινε στην Οξφόρδη να κάνει ένα ντοκτορά φιλοσοφίας μπορεί να δολοφονηθεί η δολοφονία του David δεν μας έφερε πιο κοντά στην ειρήνη. Δεν είχε απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Και όταν έλεγε ο David ότι όταν συναντούσε Παλαιστίνιους φοιτητές, οι Παλαιστίνιους που ερχόταν στο Τελαβίβ για μια συνάντηση, ήθελε να μπορεί να τους ε, αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια. Μία μέρα πριν ε, σκοτωθεί ο Ντέιβιτ μου είπε κάποιος ότι ενώ προσπαθούσα να περάσω από εκείνη την είσοδο στα κατεχόμενα ήθελε να ελέγξει τα χαρτιά μου συζήτησα λοιπόν μαζί του και όταν τελείωσε η συζήτηση αυτό που μου είπε ο άνθρωπος αυτός είναι ότι την επόμενη μέρα όταν έμαθε ότι δολοφονήθηκε ο γιος μου, λυπήθηκε πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποια βήματα έτσι ώστε αυτός ο φαύλος κύκλος βίας και θανάτου να σταματήσει. Όταν ε, έμαθα το θάνατο του γιού μου, δεν ήξερα τι θα μπορούσα να κάνω από εκεί και πέρα στη ζωή μου. Αυτό που σίγουρα ήξερα είναι ότι θα ήθελα να αποφύγω, να εμποδίσω συγγνώμη, άλλες γυναίκες να χάσουν τα παιδιά τους, να χάσουν τους γιους τους. Και ένας ιερέας ε, Εβραίος ήρθε και με βρήκε και με κάλεσε να συμμετάσχω στην ε, Ανατολική Ιερουσαλήμ σε ένα σεμινάριο με Παλαιστίνιους. Συνάντησα, θα συναντούσα εκεί και άλλους ε, γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους, άλλους συγγενείς ε, δολοφονημένων. Καταρχήν ε, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να μην πάω, όμως όταν πήγα εκεί, γιατί θεώρησα ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να καταλάβουν καλύτερα, συνειδητοποίησα ότι οι μητέρες νέων Παλαιστινίων που είχαν ε, χάσει τη ζωή τους ήταν ακριβώς την ίδια κατάσταση με μένα. Είχαν τα ίδια δάκρυα, συζητήσαμε και αποφασίσαμε από κοινού να μεταφέρουμε στον κόσμο ένα μήνυμα αισιοδοξία και ελπίδας. Το θέμα δεν είναι αν είναι κάποιος ε, υπέρ του Ισραήλ ή υπέρ της Παλαιστίνης. Πρέπει να είμαστε υπέρ της ειρήνης, πρέπει να βρεθεί λύση για να σταματήσει να δημιουργείται αυτό το μίσος μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω σε όλους να μην πάρετε θέση, αλλά να συνεισφέρετε και εσείς την εξέβρεση λύσης. Το θέμα δεν είναι η κατοχή και αν είναι κανείς υπέρ ή κατά της κατοχής. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει, λατρεύω τη χώρα μου, αλλά πρέπει να ζήσουμε σε ένα Ισραήλ με ηθικές αξίες. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να μας βοηθήσετε να πάψει να υπάρχει αυτή η κατοχή του Ισραήλ. έχουμε μια ισχυρή ομάδα γυναικών και πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει να βρεθούν γύρω από ένα τραπέζι. Κανείς δεν μας ζητάει να πολεμήσουμε είτε να διαπραγματευτούμε είτε να υπογράψουμε μια συμφωνία ειρηνευτική. Τα περισσότερα θύματα των πολέμων είναι γυναίκες και παιδιά. Θυμάμαι στο τελευταίο πόλεμο μπήκα σε ένα καταφύγιο κοντά στο σπίτι μου και εκεί ήταν μια γυναίκα με ένα μωρό νεογέννητο. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα πόσο τυχερή είμαι γιατί σκέφτηκα είμαι τυχερή γιατί έχω καταφύγιο, έχω που να πάω να κρυφτώ όταν βομβαρδίζουν την περιοχή μας. Στη λωρίδα της Γάζας όμως, μία γυναίκα η οποία μένει στο σπίτι της μπορεί να βομβαρδιστεί και να χάσει τη ζωή της από τους βομβαρδισμούς των ε, Ισραηλινών, του Ισραηλινού στρατού. Άκουσα και μια γυναίκα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Παλαιστίνης, μιλούσε για τα τρία της παιδιά, λέγοντας ότι έπρεπε να τα πάρει μαζί της και να τα οδηγήσει στο καταφύγιο. Αναρωτιόταν λοιπόν, επειδή το ένα από τα τρία της παιδιά ήταν σε αναπηρική καρέκλα, ποιον έπρεπε να πρωτοπάρει και να βοηθήσει, να κρύψει. Καταλαβαίνετε σε τι διλήμματα μπροστά βρισκόμαστε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή είναι δραματικά γεγονότα για σας. Το μέλλον όμως όλων μας όμως εξαρτάται από την επίλυση της διαφοράς σε αυτή την περιοχή. Στις 6 ελπίζω να έρθετε όλοι στην έκθεση που εγγενιάζουμε σήμερα. Είναι πολύ όμορφες εικόνες γυναικών και ανδρών πέντε από την Παλαιστίνη και πέντε από το Ισραήλ που έχασαν τους δικούς τους. Μια γυναίκα που έχασε το παιδί της, κάποιος άλλος που έχασε δύο γιους. Υπάρχει όμως και ένα μήνυμα αισιοδοξία και ελπίδας ότι μπορεί από κοινού να βρούμε λύση. Στην δυτική όχθη συνάντησα πολλές γυναίκες που κεντούν που δεν έχουν ε, χρήματα για να αγοράσουν καλής ποιότητας υλικά, κλωστή για να κετήσουν. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι η ελεημοσύνη την οποία μπορείτε να νιώσετε προς αυτούς τους ανθρώπους και να βοηθήσετε τις γυναίκες αυτές δεν είναι αυτό που χρειάζονται. Στο Τελαβίβ, στη σχολή μόδας, από κοινού με το, τη σχολή μόδας ε, Fashion School στο Λονδίνο, οργανώνουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα δυνατότητες που θέλουμε να προσφέρουμε σε γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να μπορέσουν να βρουν λύση εκτός αυτών που τους προσφέρει η περιοχή μας. Θα ήθελα λοιπόν και εσείς να βοηθήσετε. Βοηθήστε μας και εσείς. Δείξτε ότι θέλετε να βρεθεί λύση στην Μέση Ανατολή, ότι θέλετε να μας βοηθήσετε και βέβαια γυναίκες όπως η Ελέν Μίρεν, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η Μέριλ Στρίπ και η Κέιτ Μπλάντσετ θα συνεισφέρουν μαζί σας. Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Μπορώ να σας δώσω και κάποια παραδείγματα για το τι ακριβώς κάνουμε. Σκοπός του κύκλου των ε, συγγενών, των γονέων είναι να βοηθήσουμε στην συμφιλίωση και να μπορέσουμε και εμείς να συμμετάσχουμε σε κάθε προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Η διαδικασία της συμφιλίωσης ελπίζω να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκεχηρία μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε κυρία Ρόβιν Κάμελινγκ για τα λόγια σας, για την ομιλία σας που μας συγκίνησε όλους είμαι βέβαια Και είδαμε με ποιο τρόπο μερικές φορές ε, βρίσκει τη δύναμη ε, παρά το πένθος του να δώσει μάχη για κάτι που θεωρεί ότι είναι δίκαιο. Και τώρα ο κύριος Μπασά Μαραμίν. Thank Ευχαριστώ. Βλέπω πιο πολλούς Γερμενείς από ότι μέλη του κοινού. Να μιλήσω αραβικά. Όχι ακόμα. Έχουμε μόνο ευρωπαϊκές γλώσσες εδώ. Τα αραβικά δεν είναι ευρωπαϊκή γλώσσα. Όχι, όχι επίσημη. Ο Λένιν έλεγε ότι η γυναίκα που μπορεί να κρατήσει στο δεξί της χέρι ένα, μια κούνια με ένα μωρό, στο αριστερό της κρατάει το, το μέλλον του κόσμου. Εάν μορφώσει λοιπόν κανείς ε, μια γυναίκα όπως και τους άντρες, θα μορφώσει όλη την κοινωνία. Οι γυναίκες δεν περιμένουν την ελευθερία τους από τους άντρες και δεν θα έπρεπε να την περιμένουν. Θα έπρεπε να απελευθερωθούν μόνες τους και να χειραπετηθούν. Είναι δύσκολο να μεγαλώνει κανείς χωρίς ε, πρόσβαση στη μόρφωση σε περιβάλλον με ξένου ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα γιατί δεν μπορεί να ασκήσει τι θρησκευτικέ του πεπιθήσει ελεύθερα και γιατί μπορεί να περιβάλλεται από πολεμιστές όπως ε, τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Εγώ βρέθηκα περιστοιχισμένο από στατιώτες όταν ήμουν 13 και άρχισα να υψώνω την Παλαιστινιακή σημαία από τότε που ήταν έγκλημα εκείνη την περίοδο. Στα 16 μου βρήκαμε κάτι παρατημένα όπλα με και χειροβομβίδες και χρησιμοποιήσαμε τις χειροβομβίδες αυτές κατά Ισραηλινής ε, περιπολίας, περιπόλου στην ε, Χευρώνα. Τότε δεν ε, σκοτώθηκε κανείς και δεν τραυματίστηκε κανείς γιατί δεν ξέραμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν τα αφοπλήσαμε σωστά, αλλά συλληφθήκαμε. Και κάποιοι έμειναν 21 χρόνια φυλακή. 19, 17, 5, εγώ έμεινα 7 χρόνια στη φυλακή. Στη φυλακή έμαθα ότι αν γνωρίζει κανεί τον εχθρό του μπορεί να τον νικήσει ή να τον σκοτώσει. Αρκεί, ε, δεν αρκεί να τον χτυπήσει γιατί μπορεί να σκοτωθεί ο ίδιο. Επειδή μιλάει εβραϊκά, ο εχθρό μου λοιπόν έμαθα εβραϊκά και είδα μια ταινία για το ολοκαύτωμα για το οποίο δεν ήξερα τίποτα. Ε, για μα, για του Παλαιστινίου, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν το πιστεύουμε ότι συνέβη. Διότι δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό. Αγνοούμε. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αισθανθούμε συμπόνια για τον εχθρό μα. Ε, όταν δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτόν. Μετά από λίγα λεπτά από την αρχή της ταινία βρήκα τον εαυτό μου να έχει βάλει τα κλάματα. Αισθάνθηκα συμπόνια για αυτού του ανθρώπους. Ήταν πολύ δύσκολο να δω την ταινία στο τέλος, γιατί έπρεπε να ανακαλύψω αυτό το έγκλημα που έγινε και ήθελα να ε, ευχαριστηθώ την ταινία, να ευχαριστηθώ που κάποιοι δολοφονούσαν και βασάνιζαν ε, Εβραίου γιατί έχουν κάνει κατοχή στα δικά μου εδάφη, και με έχουν ε, εχμαλωτήσει. Αλλά τελικά θέλησα να μάθω περισσότερα για το ολοκαύτωμα. Το 2011, ε, πριν από πέντε χρόνια, τελείωσα το μάστερ μου ε, για το ολοκαύτωμα. Αυτό ήταν το βασικό θέμα σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ω εργαλείο για να καταλάβω τον εχθρό μου, όχι αναγκαστικά να τον ετήσω. Στη φυλακή δεν μιλάμε μεταξύ μα. Απλώ μισούμε ένα τον άλλο. Οι Παλαιστίνοι δεν χρειάζονται εκπαίδευση νομίζουμε. Ε, αλλά η εκπαίδευση είναι ένα παράθυρο. Ε, μισούμε τους Ισραηλινούς, μισούμε την ε, βία τους. Προσπαθούν να θανατώσουν την ανθρώπινη υπόστασή μας κάθε λεπτό. Πρέπει όμως να επιβιώσουμε. Ε, υπάρχει ε, στρατιωτική μάχη κατά του θανάσιμου αυτού εχθρού και εμείς είμαστε αγωνιστές. Στην περίπτωση της Παλαιστίνης, στην περίπτωση της ελευθερίας, αυτό μαθαίνουμε ότι η η ιδέα της Παλαιστίνης είναι μεγαλύτερη και πιο σημαντική από εμά το, ως άτομα. Το 92 απελευθερώθηκα μετά από 7 χρόνια στην φυλακή και έμαθα πώς να αγωνίζομαι κατά, αυτός, κατά τα, αυτού του εχθρού μόνο μετά τις σπουδέ μου. Το 94 με τη συμφωνία που έγινε αρχίσαμε να αλλάζουμε άποψη ως Παλαιστίνη. Καταλάβαμε ότι αν οι ηγέτες μας μπορούν να κάθονται και να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν τέτοιε συμφωνίε. Εγώ γιατί δεν έχω περάσει 7 χρόνια στι φυλακέ του Ισραήλ. Γιατί να σκοτωνόμαστε μεταξύ μα. Περισσότερο από 100 χρόνια προσπαθούμε να δολοφονήσουμε ένα τον άλλο. Με όποιο όπλο περνάει από τα χέρια μα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν ω τώρα. Να είναι ε, μη ασφαλεί οι Εβραίοι, οι Παλαιστίνοι να μην είναι ελεύθερη, περισσότερα θύματα και θάνατοι καθημερινά. Όταν παίξα το πρώτο μου παιδί το 1994 λοιπόν, αποφάσισα ότι ο γιο μου δεν θα πάει ποτέ σε φυλακέ του Ισραήλ και ποτέ δεν θα λιθοβοληθεί. Διότι μπορώ να τον ελέγξω, μπορώ να του εξηγήσω. Στη δική μου περίπτωση, ε, κανεί δεν το έκανε αυτό για μένα. Γιατί λοιπόν πρέπει να μιλάμε για την ειρήνη, Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μα για το δρόμο τη ειρήνη. Ε, Δυστυχώ η πραγματικότητα υπερισχύει τη ε, θεωρία. Η κατοχή συνεχίζεται, οι φρικαλαιότητες συνεχίζονται, το μίσο συνεχίζεται και η βία το ίδιο. Το 2002 ε, άκουσα στα ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, του Ισραήλ για τους αντιρρησίες συνείδησης του Ισραήλ και του Ισραηλινού στρατού. Αυτούς που δεν δέχτηκαν να κατέχουν τα εδάφια και να συμμετέχουν στο στρατό, στο στρατό αυτό που κατέχει τα εδάφια της Παλαιστίνης. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί θέλησαν να καταλάβω γιατί είναι αντιρρησίε συνείδηση το 2005. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση μαζί του τότε με τέσσερα πρώτα άτομα που προσήλθαν. Ε, φαντάζεστε τι συνάντηση ήταν αυτή μεταξύ των πραγματικών εχθρών μα που γνωριζόμαστε μισούμενο τον άλλο. Έχουμε κάνει προσπάθειε να σκοτώσουμε μεν του άλλου και από τι δύο πλευρέ. Και επί ένα χρόνο οργανώναμε συναντήσει για να καταλήξουμε να συζητάμε για ειρήνη. Το πρώτο μα ταξίδι εκτό Παλαιστίνη και Ισραήλ ήταν εδώ το 2006, σε αυτή την πόλη. Και την πρώτη χρονιά ήμασταν 300 ήδη άτομα, πρώην αγωνιστές ή φυλακισμένοι το πρώτο μα σύνθημα ήταν αυτό που είχε πει και ο Νέλσον Μαντέλα. Ότι αν θέλει να κάνει ειρήνη με τον εχθρό σου, πρέπει πρώτα απ' όλα να αρχίσει να συζητά μαζί του και μετά να γίνει ε, συνεργάτη του. Τώρα πια συνεργαζόμαστε ε, και προσπαθούμε να βρούμε λύσει. Δεν χρειάζεται να αγαπιόμαστε. Μπορούμε να συνεπάρξουμε ειρηνικά χωρί να αγαπιόμαστε, αλλά όχι να κατέχουμε ένα τον άλλο. Δυστυχώ, αν ζει κανεί στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ, ε, δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ασφαλέ το περιβάλλον. Και κάποιε φορέ, αν επιβιώσει κανεί, μπορεί να είναι τυχερό. Όχι επειδή δεν τα καταφέρνει κανεί επειδή είναι σοφό. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Δεν είναι αυτή μια φυσιολογική ζωή. Δεν μπορεί κανεί να προστατεύσει τα παιδιά του. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Το 2007, στι 16 Ιανουαρίου 2007, μετά από δύο χρόνια, αφού είχαμε οργανώσει το Combatants for Peace, ε, αγωνιστέ για την ειρήνη, ε, εγώ και τα παιδιά μου στην Ιερουσαλήμ όπου κατοικώ, Ε, βρέθηκα στο σχολείο να χάνω, ε, μπροστά στο σχολείο της να, χάνω αυτή, να κάνω τη, τη, τη δεκάχρονη κόρη μου που πυροβολήθηκε στις πόρτες του σχολείου στις 9.30 το πρωί ενώ πήγαινε στα μαθήματα ε, και έχασε τη ζωή της λίγο μετά πηγαίνοντας στον δρόμο για το νοσοκομείο. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον είναι να χάσει ένα παιδί, ιδίω ένα δεκάχρονο, που δεν ήξερε τίποτα για τον πόλεμο. Τότε ήθελα να ελπίζω ότι η Αμπίρ θα είναι το τελευταίο θύμα του πολέμου Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Δυστυχώ δεν ήταν έτσι. Αυτό που είπα είναι ότι δεν θέλω να εκδικηθώ. Θέλω δικαιοσύνη. Διότι ένα Ισραηλινό πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη μου, αλλά πάνω από 100 ε, στρατιωτέ και αξιωματικοί από το Combatants for Peace παλεύουν για τον ε, αντίθετο σκοπό και πήγαν για να αποτύσσουν φοροτιμή στο σχολείο τη, στο νεκροταφείο. Έτσι προσπαθεί κανεί να δημιουργήσει μια γέφυρα και όχι να συνεχίσει τον πόλεμο. Να δημιουργήσει μια γέφυρα για διάλογο με την άλλη πλευρά. συναντήθηκα με, 600, με μέλη 620 οικογενειών και γονεί που και αυτοί έχουν θύματα στην οικογένειά του και προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε ότι ό,τι και αν πιστεύουμε, είτε ω Ισραηλινοί είτε ω ε, Παλαιστινοί, πρέπει να μοιραστούμε αυτή τη γη. Είτε ω δύο κράτη, δύο αρχέ, πέντε κράτη, ό,τι θέλετε. Το θέμα είναι τι γίνεται με του νεκρού μα, του τάφου, τα παιδιά μα και τι οικογένειέ μα. Οι Ισραηλινοί δεν θέλουν μετά από 300 χρόνια να εγκαταλείψουν αυτό το μετά από 300 χρόνια διακριτική μεταχείριση και 3.000 χρόνια αιχμαλωσία, διακριτική μεταχείριση και σκλαβιά να εγκαταλείψουν αυτό το ασφαλέ περιβάλλον και εμεί ω Παλαιστίνοι ποτέ δεν θα εγκαταλείψουμε την ελευθερία μα. Διότι είμαστε ανθρώπινα όντα και στα χέρια μα είναι να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να πολεμάμε ή να συνεπάρχουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ραμή. Και τελευταία μας καλεσμένη, η κυρία Σουμάχερ από τη UN Women. Ευχαριστώ, Ιράτσε. Έχω έρθει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν θυμάμαι να έχω συγκινηθεί τόσο πολύ. Σας ευχαριστούμε για τις μαρτυρίες σας και τα θερμά μου συγχαρητήρια για το έργο σας. Είπατε ότι ήρθε η ώρα να καθίσουν στην τράπεζα να διαπραγματεύσουν και οι γυναίκες. Αυτά είναι πολύ σοφά Και όλα σα τα σχόλια και των δυο σα έβριθαν σοφίας και σύνεση. Και νομίζω ότι με αυτά τα σοφά υπάρχει ακόμη ελπίδα και μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την ε, κατεύθυνση. Μιλήσατε ε, για την ισότητα ε, είναι και ο Γενικός Γραμματέας εδώ και σε λίγο θα το συναντήσουμε. Πάντως σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σε αυτή την εκστρατεία. Μου είχατε ζητήσει να σας μιλήσω για το θεματολόγιο γυναίκες ε, και ειρήνη και ασφάλεια. Και συμφωνώ ότι ήρθε η ώρα να κάτσουν στην τράπεζα των Διπραγματεύσεων και οι γυναίκες. Δεν θέλω να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, γι' αυτό και θα συντομεύσω κάπως την ε, ομιλία μου για να αφήσω χρόνο για τη συζήτηση που είναι και το πιο σημαντικό. Θα σταθώ σε μερικά πράγματα μόνο. Ευελπιστώ ότι η πρωτοβουλία που μας παρουσιάσατε και το έργο σας θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες ε, τέτοιες πρωτοβουλίες ε, στην Ισραηλινή και Παλαιστινιακή κοινωνία και πραγματικά μας δίνεται ελπίδα με αυτή την πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για τις γυναίκες στην ασφάλεια και την ειρήνη. Ήδη το 2000, ξέρετε, υπογράψαμε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπαριθμό 1325. Αυτό ήταν το πρώτο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που έδωσε το σημαντικό και χειρό μήνυμα για τη σημασία που έχει η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Έκτοτε ακολούθησαν πολλά παρόμοια ψηφίσματα και πέρυσι κάναμε μια αναθεώρηση 15 χρόνια μετά το πρώτο ψήφισμα του Ηνωμένων Εθνών για το θέμα αυτό. Τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ενέκρινε το ψήφισμα 2242 που θέτει το ρόλο των γυναικών στην ασφάλεια και την ειρήνη ως βασική προτεραιότητα στο νέο πλαίσιο και τις νέες προκλήσεις παγκόσμιας ασφάλειας και ειρήνης ε, με την έξαρση της ε, βίας, ε, του προβλήματος του προσφυγικού, τον μεγάλο αριθμό των εσωτερικά εκτοπιστέντων και το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών. Είναι το μόνο ψήφισμα αυτό, το 2242, που αναγνωρίζει τις νέες προκλήσεις. το ψήφισμα επίσης ε, ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή και ηγετική θέση των γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων στην ανάπτυξη στρατηγικών προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτή η βία εις βάρος των γυναικών που διαπιστώνουμε σε πολλές κοινωνίες και μάλιστα ζητήθηκε 15% τουλάχιστον της χρηματοδότησης των ΗΠΑ και των κρατών μελών να αφιερωθούν σε θέματα ασφάλειας και ειρήνης και κυρίως σε γενικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό. Γιατί οι ομάδες και κύκλοι σαν τους δικούς σας ε, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι θα συμβάλλουμε έτσι σε μεγάλη πρόοδο. Επίσης, όταν ε, εξετάζουμε τα αριθμητικά στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι πολύ λίγες γυναίκες συμμετέχουν σε ειρηνευτικέ διαπραγματεύσεις Δυστυχώ. Και σε μία μελέτη που κάναμε στη UN Women το 1992 διαπιστώσαμε ότι από ε, ένα δείγμα 31 ε, διαπραγματευτικών διαδικασιών από το 1902 μέχρι το 2011 μόνο το 2% επικεφαλής διαπραγματεύσεων διαπραγματευτικών ομάδων, 4% ε, υπογραφών και 9% διαπραγματευτών ε, ήταν γυναίκες μόνο. Πολύ χαμηλά ποσοστά, που σημαίνει ότι με ρυθμό χελώνας προχωρούμε στην μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις διαπραγματευτικές ομάδες. Επίσης 4% μαρτύρων και υπογραφώντων. Εσείς είστε οι μάρτυρες της κατάστασης ε, και ξέρετε πως κάποια μέρα μπορεί να εδραιωθεί η ειρήνη, γιατί η δική σας συνεισφορά είναι σημαντική. Ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και άνδρες και γυναίκες θα πρέπει από κοινού και ισότιμα να συμμετέχουν σε τέτοιες ειρηνευτικές διαδικασίες. Επίσης διαπιστώνουμε ότι στις, ε, στις αστυνομίες και στους στρατούς, σε αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, η συμμετοχή των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλή, παρά το γεγονός ότι ε, έχει σημαντικό αντίκτυπο η συμμετοχή τους ε, στην ε, ευαισθητοποίηση για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Όσο περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στην αστυνομία και στο στρατό, τόσο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση θα υπάρξει για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό και θέλουμε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους και σε αυτά τα σώματα ασφαλείας. Ένα ακόμη θέμα πριν ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, το θέμα της συμφιλίωσης τη ειρηνευτική διαδικασία και της σημασία τη οικονομική χειραφέτησης των γυναικών, ώστε από τη στιγμή που συναυθεί μια ειρηνευτική συμφωνία και αποκατασταθεί η ειρήνη, θα πρέπει οι γυναίκε να θεωρούνται όχι μόνο στήματα, θύματα, αλλά και ω φορείς αλλαγής και συντελεστές της αλλαγής. Έτσι αντιμετωπίζουμε ως πραγματικούς φορείς και παράγοντες της αλλαγής και σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και τις μαρτυρίες σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Σουμάχερ. Ήρθε η ώρα για τη συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερο που ξαναβλέπουμε εκπροσώπους αυτής της οργάνωσης ε, που είναι όχι μόνο συγκινητικό το έργο της, αλλά και υποδειγματικό, είναι παράδειγμα προς Και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε από πρώτο χέρι την ιστορία, από τους πρωταγωνιστές της. Έτσι θα έχουμε και σημαντικά σημεία αναφοράς στην πολιτική μας εξέταση, αλλά ταυτόχρονα μας δίνετε και ένα μάθημα ζωής με τη μαρτυρία σας. Και είναι σημαντικό επίτευγμα ε, που ήρθατε εδώ και μας μιλάτε για το ρόλο των γυναικών στην επίλυση των συγκρούσεων. Είναι πολύ επίκαιρη και πολύ σημαντική αυτή η παρουσία. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο αξιών αυτό το ζήτημα. Δεν αφορά μόνο τη σημασία της ισότητας, της συμμετοχής των γυναικών, την ενίσχυση του παραγωγικού και χρήσιμου ρόλου της στην κοινωνία. Είναι θέμα συλλογικού συμφέροντος. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε αυτό το ταλέντο των γυναικών και τις ικανότητες των γυναικών, που είναι πάνω από το μισό πληθυσ... Ε, τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι στις διαπραγματεύσεις, στην επίλυση συγκρούσεων, στη διαμεσολάβηση, στην πρόληψη, στη διάγνωση, ε, οι γυναίκες ε, είναι πιο αποτελεσματικές και έχουν πιο ε, σημαντικό ρόλο τα συμμετέχουν και τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο θετικά όταν εξασφαλίζεται η συμμετοχή των γυναικών σε όλες αυτές τις πτυχές. Θα ήμασταν κακοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών αν δεν επιτύχουμε να αλλάξει η κατάσταση και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για δικαιοσύνη, για άσκηση και εγγύηση των δικαιωμάτων. Έχουμε μεγάλη ευθύνη στα χέρια μας. Έχουμε ευθύνη για τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη, απαραίτητο και κατεπήγον να κινητοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς ε, και όλα τα μέσα που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να υλοποιηθεί αυτή η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και όπου μπορούν οι γυναίκες να συμβάλλουν, να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο αριθμός των συγκρούσεων και των ε, ε μακροχρόνιων και των βραχυπρόθεσμων αυξάνεται δυστυχώς. Και στην Ευρώπη έχουμε περάσει κάποιου αιώνε ε, πολέμου, αλλά δυστυχώ ο κόσμο που μα περιβάλλει βρίσκεται σε συνεχή σύγκρουση. Και η διάρκεια αυτών των συγκρούσεων είναι πολύ ανησυχητική, γιατί μιλάμε για ολόκληρε γενιέ που χάνονται ή που είναι απεγνωσμένε, που δεν έχουν ελπίδα. Οπότε τόσο τα εθνικά σχέδια δράση που σίγουρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν, να ενισχύονται περιοδικά. Αλλά και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι κέρια σημασίας. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω κυρίως στο ρόλο που έχουν τα θεσμικά όργανα, προκειμένου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και οι τοπικοί φορείς, οι δήμοι, οι κοινότητες, έχουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και την επίλυση των συγκρούσεων σε μερικές περιπτώσεις είχαμε πραγματικά υποδειγματική επίλυση συγκρούσεων όταν εξασφαλίστηκε από νωρίς η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διευθέτηση αυτών των συγκρούσεων. Αυτά και σας ευχαριστώ. Εγώ ήδη έχω αγοράσει αυτά τα κορδόνια και αυτά που κέντησαν αυτές οι γυναίκες για να στηρίξω την εκστρατεία σας. Ευχαριστούμε κυρία Μπεσέρα, η κυρία Βαγένα. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Καταρχήν, ε, θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και θα ήθελα να σας εκφράσω την αλληλεγγύη μου, το σεβασμό μου και το θαυμασμό μου για το θάρρος σας ε, να αναγνωρίσετε την κατοχή των Παλαιστινιακών. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο σας. Και φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζετε καθημερινά πολλά προβλήματα. Άλλωστε βρίσκεται σχετικά στα σπάργανα αυτή η οργάνωση. Τις προάλλες ε, ακούσαμε ότι οι γυναίκες του Ισραηλινού στρατού άρχισαν να καταγγέλουν ε, καταχρήσεις που γίνονται και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Ισραηλινό στρατό στα κατεχόμενα. Οπότε φαίνεται ότι το κίνημά σας αρχίζει και επεκτείνεται και νομίζω ότι με συνεργασία των δύο κοινωνιών, Παλαιστινιακής και Ισραηλινής, ε, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Θα πρέπει να καταδικάζουμε τη βία από όποιον και διαπράτεται. Και οι πολίτες ε, ε, της Παλαιστίνης και του Ισραήλ δίνουν πραγματικά μαθήματα στις κυβερνήσεις και την Ισραηλινή, αλλά και στις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις κυβερνήσεις των υπόλοιπων χωρών τη παγκόσμια κοινότητα. Και μάλιστα αυτό που λέγατε και χθε, ε, αυτό που μας είπατε συζητήθηκε και χθε. Πού βρίσκονται οι γυναίκες στι ε, ειρηνευτικέ στις διαπραγματεύσεις. Γιατί όπως είπατε και εσείς, οι γυναίκες, ε, τα παιδιά, τα βρέφη είναι τα περισσότερα θύματα αυτών των συγκρούσεων. Οπότε βιώνουμε στο πετσί μας τις συνέπειες αλλά δεν έχουμε φωνή για να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας. Εμείς θέλουμε ειρήνη, θέλουμε διαπραγμάτευση. Εμείς το λέμε, αλλά κανένας δεν μας υπολογίζει, παρόλο που είμαστε το 50, η 51% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τι άλλο να πω, συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια, γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί έχουμε επιβδίσει πια από αυτή την κατάσταση. Είναι απάνθρωπη αυτή η κατάσταση που δυστυχώς εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το μήνυμα της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό θα πρέπει να ακούσουν οι κυβερνήσεις. Ευχαριστώ και να είστε βέβαιοι ότι έχετε την πλήρη αλληλεγγύη μας. Muy bien, pues si no hay más... Καλώς. Κυρία Αβιόρ, Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή σας σε αυτήν την ε, προσπάθεια εξέβρεσης ε, που σε καμία περίπτωση δεν αυξάνει την ασφάλεια και δεν ε, βοηθάει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε το έργο σας και βεβαίως να στηριχθείτε και από όλες τις ε, δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο μέσα από το διάλογο και στο πλησίασμα των θέσεων των εν και των δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Αλλιώς το μίσος αυξάνεται, ο τείχος που έχει οικοδομηθεί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βοηθήσουν στο να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι και τα Ηνωμένα Έθνη και όλοι όσοι πήραν θέση προς αυτή την κατεύθυνση βοηθούν στην επίλυση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και η Παλαιστινιακή Αρχή αλλά και οι αρχές του Ισραήλ να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπιόρκ και κυρία Σόιντροβα. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις αφηγήσεις σας καταρχήν αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι για ανθρώπους εγκεμένα που προέρχονται από εβραϊκές οικογένειες είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες σαν και αυτές που έχετε αναλάβει. Ότι κάνετε δηλαδή ο καθένας ένα βήμα προς τον άλλον. Πλησιάζεται ο ένας τον άλλον. Πρέπει σίγουρα μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας και να δημιουργήσουμε γέφυρες και διάλογο. Έχω την εντύπωση ότι αν οι Παλαιστίνοι με τους ε, Ισραηλινούς το καταφέρνουν, εάν βρίσκουν τρόπους να συνομιλήσουν και να πλησιάσουν οι μεν τους δε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Εγώ λοιπόν θα συνεισφέρω με όποιο τρόπο μπορώ σε αυτή τη συμφιλίωση. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Θα ήθελα όμως να αξιοποιήσω και εγώ αυτή την ευκαιρία και να σας κάνω μια ερώτηση για την παιδεία. Στη δική σας οργάνωση έχετε κάποιες δραστηριότητες που αφορούν την παιδεία, την εκπαίδευση. Γιατί είναι θεμελιώδες να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά με τις αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνουν κάποιες αλλαγές στην οτροπία, στην κοινωνία. Γιατί μερικές φορές το αγνοούμε, μια και πρόκειται για μακροπρόθεσμες πολιτικές που αποφέρουν καρπούς πολύ αργότερα. Αλλά είναι ότι το θέμα της παιδείας είναι το κέριο ζήτημα. Η σωστή διαπαιδαγώγηση με αξίες. Η οργάνωσή σας ασχολείται με τα θέματα αυτά. έχετε δραστηριότητες ε, προκειμένου να διαπαιδαγωγήσετε παιδιά με αυτές τις αξίες. Δεν μιλώ για την επίσημη παιδεία, για τις, επίσημες διάβλους ε, της εκπαίδευσης στα σχολεία, αλλά για την παιδεία που θα πρέπει να γίνεται την κουλτούρα στα παιδιά, ώστε να μεγαλώνουν αφήνοντας το μίσος ε, και τις επικρίσεις και μαθαίνοντας το σεβασμό και την συνύπαρξη. Κυρία Τζούλη. Έχω την τιμή να έχω συναντήσει τον Ρόμπι στο Ισραήλ. Τη Ρόμπι με την αντιπροσωπεία των γυναικών τον περασμένο Δεκέμβριο. Συναντηθήκαμε τότε με Παλαιστίνιες γυναίκες και Ισραηλινές. Και αναρωτιέμαι εάν μπορεί να μας μιλήσει λίγο για τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχω τεχνικά προβλήματα. Ε, πώς να μας στηρίξετε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πρώτα απ' όλα, μην πείτε ότι το μήνυμα που έκανατε σήμερα είναι απλώς ένα διαφορετικό μήνυμα από τη Μέση Ανατολή. Είναι δύο λαοί εδώ που θέλουν κάτι να πετύχουν. Την ε, επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι ο πρόεδρος Αμπάς θα είναι εδώ. Τι τέλεια ευκαιρία Είναι τεράστια ευκαιρία να ζητήσετε από τον πρόεδρο Ρίβλεν να ε, ζητήσει μια ένωση μη, οργανω... μη κυβερνητικών οργανώσεων για να υψώσουν τη φωνή τους, να σπάσει αυτό το φράγμα της σιωπής ε, και όλοι να αντιληφθούν ότι με αυτήν την οργάνωση μπορούμε να οργανώσουμε τη μελλοντική διαδικασία ειρήνευση. Οι στρατιώτε που δεν ξέρουν πώ να πουλήσουν του εαυτού του, διότι κάνουν τεράστια δουλειά, αλλά δεν ξέρουν πώ να την προβάλλουν, είναι καλό να μαθευτεί στον υπόλοιπο κόσμο αυτό. Αυτό είναι το μέλλον τη ειρηνευτική διαδικασία, τη διαδικασία συμφιλίωση. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι ένα στρατιώτη να παραδεχτεί τα κρίματά του. Ο Ισραηλινό στρατό δεν είναι χειρότερο από κανέναν άλλο. Αυτά συμβαίνουν σε όσου ε, του παρασύρει ορού τη ιστορία και πρέπει να πολεμήσουν. Βρίσκονται σε συνθήκε που είναι τελείω μη κανονικέ. Κάποιε φορέ όταν περνάω από κάποια checkpoint και κοιτάζω τους στρατιώτες ε, στις με τις στολές τους, είναι τόσο νεαροί που είναι σαν παιδιά, σαν παιδιά μου τους βλέπω. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να τους δίνουμε στα χέρια τους, πώς μπορούμε να τους βάζουμε σε αυτή την τραυματική εμπειρία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, να πρέπει να λάβουν αποφάσεις που ε, θα είναι τόσο σοβαρέ για το αν κάποιο πρέπει να περάσει από το checkpoint ή όχι, αν έχει άδεια. Και κάποια γυναίκα που θα ζητήσει να περάσει στο σημείο αυτό ελέγχου μπορεί να έχει το μωρό τη από την άλλη μεριά και το μωρό να πεθάνει αν δεν ε, περάσει. Και δεν νομίζω ότι αυτοί οι γονεί αυτών των ανθρώπων που στέλνουν ε, στο στρατό λέγοντα σκοτώστε την Παλαιστίνα, ε, βρείτε μπροστά σα. Κανονικοί άνθρωποι είναι από κανονικέ οικογένειε. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Και τι να πει αυτό στο σπίτι του, στου γονεί του. Δεν μπορεί να του πει τι είδε. Και καμιά φορά έρχεται να μα μιλήσει εμά ο στρατιώτη. Όμω Πολλέ φορέ μπορεί να πάρει στα χέρια του το όπλο του πατέρα του, να πάει να μεθύσει και τελικά να τραυματίσει κάποιον από ατύχημα. Ε, αυτό συμβαίνει κάποιε φορέ. Αυτά είναι τα ε, τραγικά γεγονότα. Υπάρχει πιο ενδοκογενειακή βία από ό,τι είχαμε ποτέ και περισσότερη βία στα σχολεία. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Καμία χώρα δεν μπορεί να κατέχει μια άλλη για περίπου 50 χρόνια και να μην περιμένει ότι αυτό θα ε, επηρεάσει τον ηθικό ιστό τη κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε από αυτά. Πρέπει να μάθουμε πώς θα επηρεάσουμε τη σκέψη των ανθρώπων και τα συναισθήματά τους. Μπορεί κανείς να ενημερώσει, να ασκήσει πίεση, να μιλήσει στους ελληνούς τα κατεχόμενα. Αυτό είναι η καλύτερη στήριξη που μπορείτε να μας δώσετε. Ρωτήσατε και το συζητήσαμε και το πρωί για μια ιδέα που είχαμε. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που έρχονται από το Λεβάντε, δηλαδή Μαρόκο, οι Εβραίες γυναίκες που από το Μαρόκο, την Τινησία, την Αλγερία, τις χώρες της Βορειοαφρικής. Και ζουν σε πολύ μικρές πόλεις γύρω από το Ισραήλ. Δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίε και συνήθως ψηφίζουν προς τα δεξιά. Πώς να τις πλησιάσουμε, διότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Αυτές τις γυναίκες θέλουμε μαζί μας και με αυτές θέλουμε να μιλάμε. Εάν μπορούσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Δεν μιλάω τώρα για λεφτά, γιατί είναι βρώμικο το χρήμα. Αλλά αν μπορούσαμε να πάμε και να μιλήσουμε σε αυτές τις γυναίκες, θα σας φαίνεται τρελό, αλλά το κάναμε, το κάναμε με μια ομάδα. Παλαιστίνιες και Ισραηλινές γυναίκες. Μαγειρέψαμε, μαγειρεύαμε μαζί συστηματικά επί ένα χρόνο, φτιάχνοντας γεύματα με μαρμελάδες και ε, τουρσιά. Ε, εδώ αυτό που καταφέραμε είναι να ακούσουμε τις ιστορίες η μια της άλλης, να καταλάβουμε ποιες είμαστε, από πού προερχόμαστε και πώς βλέπουμε τα πράγματα, πώς βλέπουμε όλη μας την ιστορία, ποιες είναι αυτές οι γυναίκες. Ε, τέτοια συνενοχή δημιουργήθηκε μεταξύ μας, τέτοια ομοψυχία που σκεφτήκαμε ότι αυτό που είδαμε είναι ότι οι γυναίκε που έρχονται από αυτέ τι χώρε ξέρουν να μαγειρεύουν πολύ καλύτερα από τι γυναίκε που είναι σκενάζοι, που έρχονται από την Ευρώπη, δηλαδή οι Εβραίε που έρχονται από την Ευρώπη. Καταλάβαμε ότι μπορούμε να πάμε και να μαγειρέψουμε και στον κύκλο που κάνουμε γύρω από τη φωτιά καθόμαστε και λέμε ιστορίε. Και ε, αυτό ένα από τα προγράμματα που έχουμε λέγεται Ιστορία από την ανθρώπινη σκοπιά. ιστορία through the Μιλάμε με 17 χρόνια αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Πριν πάνε στρατό. Και όσο πιο πολύ τους μιλάμε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Είναι πολύ πιο σημαντικό να τους εκπαιδεύσουμε ε, αυτούς αντί να περιμένουμε τους ενηλίκους. Δεν θα περιμένουμε να μεγαλώσουν τα τρίχρονα βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε τέτοια μορφωτικά προγράμματα και για ενηλίκους και για εφήβους το μουσείο του ολοκαυτώματος ας πούμε, όχι για να συγκρίνουμε ποιος υπέφερε πιο πολύ, αλλά αν δεν καταλαβαίνει κανείς το φόβο, το φόβο που είναι μέρος του γενετικού υλικού των ε, Εβραίων, του, λαού, του, του εβραϊκού λαού, δεν μπορεί να καταλάβει πώς να διαμαρτευτεί και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς αισθάνεται μια γυναίκα για το χωριό τη, για το χωριό που μπορεί να καταστράφηκε το 1948 και τώρα είναι μέρος του Ισραήλ. Ε, η Παλαιστίνια που βλέπει το πηγάδι που παίρνει νερό να είναι ένα πηγάδι που παίρνει νερό ένα παιδί μια άλλη γυναίκα. Ε, όλα αυτά τα θέματα είναι θέμα εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. και ε, το Πανεπιστήμιο Georgetown μας από την Washington μα συμβούλεψε και δημιούργησε ένα άλλο πρόγραμμα ιστορία από την ανθρώπινη σκοπιά για πολλά επαγγέλματα, για καλλιτέχνες, για δασκάλους και καθηγητές ένας τρόπος ο καθένας να καταλάβει τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι ε, αρχίζουμε να καπιόμαστε ξαφνικά και τρώμε μαζί χούμους. Σημαίνει ότι αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα ένα τον άλλο. Αυτό επιτρέπει να έχει κανείς ενσυναίσθηση συνέστηση για την ε, προοπτική του άλλου και είναι το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε ε, να γίνει και να πετύχει. Μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια να του μορφώσουμε και να του εκπαιδεύσουμε όλου. Αλλά πραγματικά θυμώνω όταν μου λένε ότι οι Παλαιστίνοι ε, μαθαίνουν στα παιδιά του να μισούν. Σα διαβεβαιώ, εάν είχα μεγαλώσει σε καταβλισμό προσφύγων, δεν θα χρειαζόμουν κανένα κύκλο μαθημάτων να μου μάθει το μίσο. Ε, είναι απλό. Ας δούμε τις μητέρες αυτών των 14χρονων ε, που βγαίνουν με μαχαίρια και να σκεφτούμε αυτές τις μητέρες που μπορούμε να τις βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα των παιδιών τους να... και την πιθανότητα τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν βίαιη συμπεριφορά. Θα πρέπει να τις πλησιάσουμε και μέσα από τα σχολεία. Αυτό μπορείτε να κάνετε για να μας στηρίξετε. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι ένα τετράχρονο αγόρι, ένα εντεκάχρονο παιδί που δεν έχουν καμία ευκαιρία στη ζωή του. Δεν είναι το δικό μου 14χρονο εγγόνι που μπορεί να πάει όπου θέλει, να παίξει μπάσκετ όπου θέλει, να κάνει κολύμπι και να πάει σε ένα σχολείο με δημοκρατικές πεπιθήσει. Αν είμαι 14χρονο Παλαιστίνιο, μάλλον μετά το σχολείο δεν έχω τίποτα να κάνω και μάλλον θα θέλω να μιμηθώ τον πατέρα μου που ήταν μέρο τη δεύτερη ηττιφάδα και ήταν ήρωα. και μπορεί να μην καταλαβαίνω ότι δεν είμαι άτρωτος, να αισθάνομαι αίτητος και εάν ε, δεν ε, έχω τέτοια συνέστηση δεν θα καταλάβω ότι μπορώ να σκοτωθώ. Πώς θα τα μορφώσουμε αυτά τα παιδιά. Νομίζω, παιδεύοντας τις μητεράδες τους, δεν λέω ότι είμαι κατά της εκπαίδευσης ε, των παιδιών των ίδιων. Φυσικά και όχι. Οργανώσαμε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση για τέτοια ξεστρατισμένα παιδιά. Και είδαμε στην αρχή ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά Ισραηλινών και Παλαιστινίων σιγά σιγά κατανοούν ότι είναι ολόιδια. Ακούνε την ίδια μουσική, τρώνε το ίδια φαγητά, διασκεδάζουν τα ίδια πράγματα. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα του Ισραήλ και τη Παλαιστίνη. Εάν ρωτήσει κανεί τον οποιοδήποτε 17χρονο στο Ισραήλ, αν έχει ε, συναντήσει Παλαιστίνιο, θα σα πει όχι. Ίσως σε μια τάξη των 35 ατόμων να έχει βρεθεί και ένα Παλαιστίνιο. Αλλά γιατί, γιατί άμα πάω σε μια τάξη σε Παλαιστινιακό σχολείο με κοιτάνε. Γιατί να σκεφτούν ότι διαφέρω από τους... Ε, από τους ε, στρατιώτες που έχουν συναντήσει του Ισραήλ ή από τους ε, καταπατητές των εδαφών τους. Εδώ Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από αυτή την προσπαθεια προσεγγισης προσέγγιση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Σίγουρα χρειαζόμαστε και κονδύλια, αλλά πάρα πολλά χρειαζόμαστε υποστήριξη, υποστήριξη για να μιλήσουμε σε όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάποια αλλαγή, κάποια διαφορά. Να ασκήσουμε πίεση για να γίνει αυτή η αλλαγή, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τη διαδικασία συμφιλίωσης. Ακόμα και να οργανωθεί εδώ μια συνδιάσκεψη για τη συμφιλίωση, προτείναμε σήμερα το πρωί. Να το οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσκληθούν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με διαδικασίε συμφιλίωση σε όλο τον κόσμο και να δημιουργηθεί ένα πραγματικό πλαίσιο γι' αυτό. Και άνθρωποι που έχουν ζήσει προσωπικά διαδικασίες συμφιλίωσης για να γίνει αυτή η ριζοσπαστική κίνηση, αυτή η καμπή σε συναισθηματικό επίπεδο. Μιλήστε μαζί μας. Αυτό είναι το βασικό. I just want to say κανείς να τους πει αγαπήστε τους στρατιώτες που σας ταλαιπωρούν, που σας περνούν μέσα από τα checkpoints, τους οποίους βλέπουν σαν εχθρούς. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήρθατε στη συνεδρίασή μας, που μοιραστήκατε μαζί μας την προσωπική σας εμπειρία τα προσωπικά σας βιώματα και σας ευχαριστώ θερμά για το τεράστιο έργο που κάνει αυτή η οργάνωση, η μη κυβερνητική οργάνωσή σας, το Parent Circle και νομίζω ότι καταλάβατε και από τα σχόλιά μας πόσο συμπάσχουμε μαζί σας και πόσο αλληλέγγυοι νιώθουμε. Μακάρι να βρεθούμε κάπου στο δρόμο και μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, να σημειωθεί πρόοδος και να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος της ε, συμφιλίωσης και της ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Πάντως, ε, να είστε βέβαιοι ότι τα μέλη της Επιτροπής μας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουμε οργανώσεις τις δικές σας για να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους ε, προς το κοινό συμφέρον και προς τους κοινούς αυτούς στόχους. Σας ευχαριστώ θερμά. περαιώσαμε το σημείο αυτό της ημέρησης διάταξης. Αν δεν έχουμε τίποτα για τα διάφορα, να σας υπενθυμίσω ότι 16 Ιουνίου θα είναι η επόμενη μας συνεδρίαση, μεθαύριο δηλαδή ουσιαστικά. 9 με 10 το πρωί πρόκειται για κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Απασχόλησης στα πλαίσια ε, της κοινή μας προσπάθειας για το συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και εξέταση των σχετικών τροπολογιών. Όσοι πιστοί προσέλθετε.